Okay, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε με την έκτακτη αυτή συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Συνήθως δεν είμαι και πολύ υπέρ τέτοιων έκτακτων συνεδριάσεων, αλλά δεδομένου ότι έχουν μαζευτεί διάφορα ε, ζητήματα από τριμερείς διαλόγους, έπρεπε να συνεδριάσουμε. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν επιθυμίες να τροποποιηθεί κάτι, παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου. Θα ήθελα οι δύο ψηφορίες, οι 10 και οι 11, για το Μαρόκο να τις αναβάλουμε, να τις αναφέρουμε τη μέση διάταξη. Ωραία. Για το 10 και το 11 λέτε, έτσι. Να αφαιρεθούν από την ημερήσια διάταξη πρέπει να το ζητήσουν οι τρεις ε, βουλευτές ή μια πολιτική ομάδα. Λοιπόν, μετράω. Εντάξει. Και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε το αίτημα αυτό. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ της αναβολής. Ας το κάνουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε το αίτημα. Συνεπώς παραμένει στην ημερήσια διάταξη. Κάτι άλλο για τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη. Όχι από ό,τι βλέπω. Ωραία. Σημείο 2. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες που χρειαζόμαστε. Και περνάμε στην πρώτη ψηφοφορία. Πρόκειται για την ε, προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη της Γενέβης, της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της περίφημες. Μία ψηφοφορία μόνο, Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε με ομοφωνία. Συγχαρητήρια κύριε Μπεγκίν. Και περνάμε σε ένα άλλο συνδεδεμένο με αυτό θέμα, που είναι η δεύτερη έκθεση που θα ψηφίσουμε. Εδώ έχουμε αρκετές τροπολογίες. Και αρχίζουμε με την τροπολογία αριθμός 7. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αριθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για τροπολογία αριθμός 5. Τέλος. Και απορρίφθηκε, σαφώς. Και αριθμός 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε ομόφωνα. Συγχαρητήρια κύριε Χάντζεν. Συνεχίζουμε. Περνάμε στο σημείο 5 τώρα. Πρόκειται για προφορική ερώτηση για μέτρα αντι-dumping της Κολομβίας. Με μία ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Σαφώς. Σημείο 6. είναι το αποτέλεσμα τριμερούς διαλόγου για το πλαίσιο ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων. Θα δώσω το λόγο βέβαια στον εισηγητή μας, τον κύριο Προύστα, αλλά πρώτα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Και εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Ο κύριος Προύστ. Παρακαλώ κύριε Προύστ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα και εσάς, Πρόεδρε της Επιτροπής ΙΝΤΑ, για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγατε τους τριμερείς διαλόγους από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλευρό μας. Είμαι ήταν συγητής και ο κύριος Μπάτι Κόφερ, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ για να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα αυτό και ευχαριστώ και όλους τους κοιόδη συγητέ, που και αυτοί από κοινού δούλεψαν υπέρ του γενικού συμφέροντο πάντα. Και αν καταφέραμε στο θέμα αυτό να προχωρήσουμε γρήγορα, <clears throat> γιατί όντω πίεζε η κατάσταση, το θέλανε και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μας, εγώ πάντα λέω ότι είναι και το τρίτο σκέλος του τέλους της αθότητας στην Ευρώπη μετά από το CFDI και άλλα μέτρα που υιοθετήσαμε, τώρα νομίζω ότι είναι καλύτερα εξοπλισμένη η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει σήμερα την παγκοσμιοποίηση. Πάντα ήμασταν υπέρ της ποιότητας της εργασίας μας. Ακόμα και αν προχωρήσαμε γρήγορα, δεν θυσιάσαμε την ποιότητα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας και ελπίζω η σημερινή ψηφοφορία να γίνει πιο συγκεκριμένη το Φεβρουάριο στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ πάντως όλους για τη βοήθειά σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Προύστ. Προύστ, καλά δεν το είπα, λέει ο πρόεδρος. Μεγάλη επιτυχία αυτή. Τη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημείο 7. Και εδώ είναι μια άλλη επιτυχία σε τριμερή διάλογο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα οριζόντια μέτρα. Πάλι μία ψηφοφορία και γι' αυτό. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας επίσης εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου. Ο κύριος Χέλνερ, ο εισηγητής μας, δεν είναι εδώ. Συγχαρητήρια πάντως. Σημείο 8. Τρίτος τριμερής διάλογος, τον οποίο ολοκληρώνουμε σήμερα με αυτή την ψηφοφορία. Πολλή δουλειά κάναμε τους τελευταίους μήνες. Κάθε εβδομάδα είχαμε τριμερείς διαλόγους. Και για μένα ήταν δύσκολοι αυτοί οι μήνες. Έχει να κάνει με το Brexit, με την ομοθεσία για το Brexit. Και εμείς πρέπει να ψηφίσουμε για την κατανομή των δεσμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ μετά την αποχώρηση του Βασιλείου. Μακάρι να μην γίνει βέβαια, έτσι. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς ποιο θα είναι το τέλος αυτής της ιστορίας. Με μία ενιαία ψηφοφορία ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίθηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ την εισηγητριά μας, την κυρία Κουίστφατ Πρόβολ. Άρα ολοκληρώσαμε τρεις τριμερείς διαλόγους. Μπράβο μας. Επόμενο σημείο. Nine, uh, the uh, agreement in form of exchange of letters between the... Πρόκειται για ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε σχέση με τη διαδικασία επίλυση διαφορών του ΠΟΕ. Μία ψηφοφορία και εδώ ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με σαφή πλειοψηφία. Συγχαρητήρια Λούλιο. Και τώρα ερχόμαστε στο σημείο 10. Εδώ έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις πριν αρχίσουμε με τα σημεία 10 και 11. Την πέμπτη που μας πέρασε πήρα επιστολή από τον Επίτροπο Μοσκοβισή που περιλαμβάνει την ανταλλαγή της DigiTaxi και του πρέσβη του Μαρόκου για την βελτίωση της ανεχνησιμότητας των προϊόντων που μας έρχονται από τη Δυτική Σαχάρα. Εμείς ζητήσαμε ένα τέτοιο μηχανισμό σε Επιτροπή και συνεπώς την επιστολή αυτή και το παράρτημα το στέλνω στους συντονιστές ερωτώντας κατά πόσο αυτό μας αρκεί για να δώσουμε την ε, σύμφωνη γνώμη μας, για να ψηφίσουμε και να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη. Η μεγάλη πλειοψηφία των συντονιστών απάντησε ότι ναι, αρκεί και μπορούμε να ψηφίσουμε. Εξού και μπήκε στην ημερήσια διάταξη για ψηφοφορία αυτό το θέμα. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερο, έγινε συζήτηση για την ε, ανεξαρτησία της εισηγήτριας. Είναι θέμα αρμοδιότητάς μου και θα υπάρξει διερεύνηση από Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμως η κυρία Λαλόντο δεν θέλει να έχει πλέον την ευθύνη για αυτό το θέμα. Οπότε ανέλαβε άλλος την αρμοδιότητα. Ο κύριος Ζαντό, από πλευρά των Πρασίνων ζητήσαμε μαζί με τους σοσιαλιστές να μην ψηφίσουμε, γιατί θεωρούμε ότι το γεγονό ότι η κυρία Λαλόντα αποσύρθηκε, δεν αναλαμβάνει πια αυτή την έκθεση, επειδή φαίνεται ότι υπάρχει κατάφορη σύγκρουση συμφερόντων και το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει η κυρία Λαλέντη είναι αυτό, αλλά η έκθεση αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων. Και επειδή δεν έχει αλλάξει ούτε κόμμα στην έκθεση, εμεί θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή αποτελεί καρπό και αποτέλεσμα μια σύγκρουση συμφερόντων και από πλευρά των πρασίνων, με τι άλλο, δεν θα συμμετάσχουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε. Δεν βλέπω να ζητάει κανεί άλλο το λόγο. Οπότε θα ψηφίσουμε. Ξεκινάμε την 61 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 64, ε, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά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 Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 συμβαστική υπέρ. Ζητώ συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, ξεχάσαμε την 111. 111 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά Ζητώ συγγνώμη. Ξεχάσαμε επίσης την 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε. Νομίζω ότι εγκρίθηκε 131 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Τρεις ταυτόσημες 132, 133 και 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Η 8 εγκρίθηκε 134 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 145 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 146 σε δύο τμήματα. Το δεύτερο καταπίπτει. Ψηφίζουμε το πρώτο. Το πρώτο τμήμα του 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 136 υπέρ. Α, καταπέπτει, συγγνώμη. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 157 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. 160-161 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 162 υπέρ. Με ηρεμία. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 168 υπέρ. Τώρα έχεις δίκιο. Ξέχασα την συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 169. 170 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 12 αρχή της ψηφοφορίας τέλος Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Α, ελέγχουμε την 17. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τριάντα έξι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 επτά υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή, 47 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ελέγχουμε αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. 56 καταπίπτει, 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1 υπέρ, 2 αποχές, απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Αρχή της ψηφοφορίας για τη δύο. Τέλος. Εγκρίνεται. Τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα Ψηφίζουμε όσον αφορά την γνωμοδότηση αγκριένα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 6 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά νομίζω ότι εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Το δεύτερο τμήμα του Άγκρι 6. Τέλος, εγκρίνεται Άγκρι 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην αλία. Τροπολογίε Αλία. Uh, uh, Τροπολογία 3, υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, Αποχέ. απορρίπτεται. Άφετ, 1 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Άφετ 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται άφετ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άφετ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άφετ 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άφετ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Άφετ 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 πρώτη πρόταση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα το ψήφισμα στο σύνολό του άρχεται η ψήφος ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται με 24 υπέρ. Συγχαρητήρια. Στην κυρία Χάκη. Πάμε στο σημείο της μερικής διάταξης 11. Έχουμε την πρώτη προλογή, την 5, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται την τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται και τρεις τροπολογίες που είναι ταυτόσμες, η 3, η 4 και η 6, υπέρ, κατά, αποχές, απόρριπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, Άρχεται η ψηφοφορία για την 3, 4 και 6. Τέλος ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Και ψηφίσουμε ολοκληρωτικά για το σύνολο της πρότασης. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Good live. Εγκρίθηκε η πρόταση σου για τις ποσοστώσεις. Χαρητήρια. Το σημείο 12 είναι υπόλοιπα θέματα. Δεν υπάρχει κάτι από την πλευρά μου. επόμενη συνεδρία είναι στις, 23, στις 3 Ιανουαρίου. Καλό διάλειμμα για τις διακοπές Χριστουγέννων. Γεια σας.